Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε μετά από το διάλειμμα που κάναμε όλοι, εκτός από αυτούς που ήμασταν εδώ και συζητούσαμε για την αποστολή για την Τσεχία. Τώρα θα περάσουμε στην απαλλαγή του 2008, το 8ο σημείο της ημερησίας διάταξης για τα άλλα θεσμικά όργανα και ξεκινάμε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ελπίζω να έχετε όλη τη σωστή λίστα ψηφοφοριών. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Είχα ετοιμάσει για δύο ώρες την ομιλία μου, οπότε καθίστε, ησυχάστε, γιατί έχω πολλά σημαντικά πράγματα να πω. Όχι, πλάκα κάνω. Ε, να ψηφίσουμε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είστε έτοιμοι. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Συνεχίζω στα αγγλικά. Θα είναι πιο εύκολο. Ξεκινάμε λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση απόφαση στο σύνολό τη με την τροποποίηση. Μπορείτε να ψηφίσετε. Κάποιος ψάχνει την κάρτα του ακόμα. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 3 κατά. Καμία αποχή. Και περνάμε τώρα στο ψήφισμα. Αιτιολογική σκέψη Α, τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έξι. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. The vote is closed. It's Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Εδώ έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία, όπως ζήτησε το ΕΛΚ. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Α, να ελέγξουμε και πάλι. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 12-11. Τροπολογία αριθμός 10 τώρα. Υπέρ. Κατά. Κατά είναι οι σοσιαλιστές. <laughs> Sorry, Maria. <laughs> It's okay. It's rejected. <laughs> Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται νομίζω. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 13 ψήφοι υπέρ. 16 τώρα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 21. Εδώ έχουμε δύο τμήματα. Το ΕΛΚ το ζήτησε. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Με προφορική τροποποίηση για τις προθεσμίες. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 22, τροπολογία 22, ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 12 ψήφι υπέρ. 23 τώρα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24. Εδώ έχουμε τρία τμήματα. Ζήτησε κατά ψηφοφορία ε, η ομάδα των σοσιαλιστών. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, απορρίπτεται, διορθώνει πρόεδρος. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25. Who is in υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε το τρίτο τμήμα. Καλώς. Θα ελέγξουμε το τρίτο τμήμα, οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το τρίτο τμήμα. Τέλος της φοφορίας. Εγκρίθηκε. 13, 11. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική αριθμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 τώρα τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές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 απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ναι, θα ελέγξουμε. Καλά, αν λέτε να ελέγξουμε, θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 43. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Με μία ψήφο διαφορά. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε. Τέλος της προφορίας. Απορρίφθηκε. Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Α, ξέχασα τις 47 λέει η Πρόεδρος. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται, διορθώνει ο Πρόεδρος. Αφετ 1. Υπέρ. Κατά. Ωραία. Ψηφίζουμε unblock. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί. Μέχρι την 8. Αφετ 8. Όλες μαζί. Ναι ή όχι. Μέχρι την έξι. Τις πρώτες τρεις. Ωραία, πρώτες τρεις λοιπόν μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ωραία. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αφέτ 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αφέτ 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αφέτ 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αφέτ 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αφέτ 9 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 12-11 το αποτέλεσμα. Ωραία. Τώρα ονομαστική ψηφοφορία για ολόκληρο το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. 21 ψήφι υπέρ, 3 κατά. Συγχαρητήρια. Και τώρα θα περάσουμε στο 9. Απαλλαγή 2018. Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Λοιπόν, ξεκινούμε από την ψηφοφορία για την παράγραφο 1, τροπολογία 1 και 2. Υπέρ, κατά, τροπολογίες, ε, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία σε ό,τι αφορά την πρόταση απόφαση στο σύνολό τη όπω τροποποιήθηκε υπέρ Αν θέλουμε να αναβληθεί είναι συν. Αν δεν θέλουμε να αναβληθεί είναι πλην. Έτσι δεν είναι. Όχι. Ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή, για την αναβολή. Οπότε συν. Βάλτε ένα συν σας παρακαλώ. A roll call vote. We have one and two and then we have the roll call vote. Έχουμε την 1, την 2, μετά την ονομαστική ψηφοφορία και μετά την 3. Και μετά ολοκληρώνει η ψηφοφορία. Έτσι ώστε όλοι να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. 23 ψήφοι υπέρ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και τώρα πάμε στο ψήφισμα. Τροπολογία υπαριθμών 3. Ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 16 πέρε 7 κατά μία αποχή. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, 7 κατά και μία αποχή. 27. Καταπίπτει. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε αυτό. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 14 υπέρ, 10 κατά, καμία αποχή, 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Όχι, συγγνώμη. 30, έτσι. Ναι, εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα έχουμε την 15 τμήματικά το πρώτο, το πρώτο τμήμα έχει αποσυρθεί οπότε ψηφίζουμε μόνο, μόνο στο δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να το επαληθεύσουμε βεβαίως άρχεται η ψηφοφορία για την 36 τροπολογία 36 μια στιγμή πέρας ψηφοφορίας Ευχαριστώ Μάρκους. Απορρίπτεται σαφώς 6 υπέρ 18 κατά καμία αποχή. 37. Όχι δεν καταπίπτει. 37 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα περνάμε στις τροπολογίες ε, της Επιτροπής Συνταγματικών Ζητημάτων. Αύκο 1 ε, μάλλον 3 και 4 να τις δούμε από κοινού, τροπολογίες 3 και 4 από κοινού, υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 6 και 7 από κοινού, υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνονται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του ψηφίσματος, το σύνολό του, επί του συνόλου μάλλον όπω τροποποιήθηκε, υπέρ όχι, είναι ονομαστική ψηφοφορία, οπότε άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 23 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή, συγχαρητήρια. Και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη απαλλαγή για το, Ευρω... για το ελεγκτικό συνέδριο. Ψηφίζουμε πρώτα επί του συνόλου Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 24. Σπάνιο αυτό. 24 ψήφου υπέρ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 11 τμηματικά. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε αυτό παρακαλώ. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 11. Υπερψηφίστηκε με μία ψήφο. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Μόλις ψηφίσαμε το 13 όμως. 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 16 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 17 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 18 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε παρακαλώ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 12-11 εγκρίνεται. Ο κύριος Κούς είναι υπεύθυνο. Λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. 22 υπέρ. Πολύ ωραία. Και περνάμε τώρα στο ε, δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης απόφασης επί του συνόλου υπέρ, μάλλον ψηφίζουμε πιο συγκεκριμένα, άρχεται ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, ...22 υπέρ, 2 κατά. Τροπολογία 1. Συγγνώμη, τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε αν θέλετε.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 Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε βεβαίως. Κανένα πρόβλημα. It's rejected. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 τμηματικά Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ναι, πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό. Έχουμε μια ψήφο παραπάνω. Ο κ. Τσανεύσκη θα έχει την αποφασιστική πτήση ψήφο. Άρχεται η ψηφοφορία ε, για το δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 20. πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 13-12 ατύχησε στόμας Συγγνώμη, έχουμε και την 21. Ξέχασα την Ολυβία και τη Ραμόνα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στη Γιούρι. Η τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. Γιούρι 7. Γιούρι 7. Αμπλόκ 7, 8, 9. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12-13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Γιούρι 15 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά πρώτο ή δεύτερο τμήμα λάθος έκανε πρόεδρος αντί για κατά είπε δεύτερο τμήμα first, του πρώτου τμήματος, λοιπόν. Κατά του πρώτου τμήματος. Μικρή διαφορά, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρινέται. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Close Πέρας. 21 υπέρ, 3 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια. Πάμε στο τμήμα 6, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Εκεί έχουμε την τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά ακολουθεί η ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση απόφαση του συνολό της όπως τροποποιήθηκε πρέπει να ψηφίσουμε αν θέλετε αναβολή πρέπει να ψηφίσετε συν εάν δεν θέλετε αναβολή πρέπει να ψηφίσετε μείον κατά δηλαδή άρχεται η ψηφοφορία αναβολή είναι το συν και μία αναβολή είναι το μείον, του πλήν. Πέρας ψηφοφορίας 24 συν μία αποχή. Έχουμε λοιπόν μια τροπολογία στην πρόταση ψηφίσματος αριθμός 2. οποίος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική ψηφοφορία, αίτημα των σοσιαλιστών. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 4. Πέρας παρακαλώ. 16 υπέρ 8 κατά εγκρινέται χωρίς αποχές. Τροπολογία 5. Ονομαστική ψηφοφορία και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ 10 κατά και μία αποχή. Τροπολογία 6, πρώτο τμήμα από τα δύο. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Σοσιαλιστές εποχή. First part. Το πρώτο τμήμα έχει αποσυρθεί. Έτσι λένε οι σοσιαλιστές. Το πρώτο τμήμα έχει αποσυρθεί. Είναι δική του η τροπολογία. Δεύτερο τμήμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα δείξουμε ευελιξία. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε μία ψηφοφορία δύο τμήματων για την 16 υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 προς 11 χωρίς αποχές. 14. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ ονομαστική ψηφοφορία μετά τα των σοσιαλιστών άρχεται η ψηφοφορία πέρας 24 υπέρ. Μία αποχή. Κανέν, καμία ψήφος κατά. Στο Βρετανικό Συμβούλιο, όπως το λένε, δεν nose have it, Λοιπόν, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25, συγγνώμη, προηγούμενα ήταν 24. 25 έχουμε μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία της 25, δεν υπάρχει. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Καταπίπτει. Είναι λάθος η οδηγία εδώ η παρατήρηση. Οπότε πρέπει να ψηφίσουμε την τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 ονομαστική ψηφοφορία μετά από ετοιμότητα των σοσιαλιστών άρχεται η ψηφοφορία πέρας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 Έχουμε ένα πρώτο τμήμα με μια προφορική τροπολογία, fully regrets. Υπάρχει κάποια ένσταση. Όχι. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, strictly and in fully transparency. Υπάρχει κάποια ένσταση για το δεύτερο τμήμα της προφορικής τροπολογίας αυτή. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 39 δύο τμήματα ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 να ελέγξουμε λέει για το δεύτερο τμήμα της 39 Έχετε την ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 13 προς 12. Ήταν μικρή η διαφορά. 41 υπέρ. Όχι, έχουμε μια αποχή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42-43 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνονται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ονομαστική ψηφοφορία για την 52 άρχεται η ψηφοφορία πέρας είναι 24 υπέρ, 0 κατά και μία αποχή. 54 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Οι επόμενες τρεις. Έχετε τις ίδιες θέσεις και τις επόμενες τρεις. Ωραία. 55, 56, 57 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε την 58 Να ζητάτε έλεγχο τα μέλη, αν θέλετε. It's 19 to 6. 19 έναντι 6. Ήταν σαφής η διαφορά. 60. 60 και 61 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 62 έως και 64 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται συνολική ψηφοφορία ονομαστική για το σύνολο του πρώτα ψηφίσματος άρχεται ψηφοφορία όπως τροποποιήθηκε εναντί μία. Συγχαρητήρια. Πάμε στην Επιτροπή των Περιφερειών. Υπάρχει μια τροπολογία 1 για αναβολή. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Σοσιαλιστές. Κατά. Ποιος θέλει να πόσχει, Κανείς. Οπότε απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα ψηφίζουμε ονομαστικά για να χορηγήσουμε την απαλλαγή. Χορηγούμε την απαλλαγή διότι έχουμε ψηφίσει κατά στην τροπολογία 1 του κυρίου Πέξα. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Χορηγείται λοιπόν η απαλλαγή, εγκρίνεται 18 έναντι 7 και 0 αποχές.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 αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά να ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 έως και 14 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί ναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ελέγχουμε την 16 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 12 με 12 και μία αποχή 17 υπέρ κατά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 αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ 2 κατά, μία αποχή. Πάμε. Τώρα στον Ευρωπαίο Συνήγορο του Πολίτη, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Και έχουμε πρώτα ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση απόφασης να δοθεί η απαλλαγή. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. 23 υπέρ, ένας κατά, καμία αποχή. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 12-11 και μία αποχή. 3. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ για την τρία. Ξανά. Ποιο είναι υπέρ τη τρία. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέντε. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έξι. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οχτώ. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εννέα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 Πέρας της ψηφοφορίας. 23 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Περνάμε στο τμήμα 9, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Πρώτα ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση απόφαση στο σύνολό της. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Η 22 υπέρ, κανένας κατά καμία αποχή. Τροπολογία αριθμός 1 τώρα. Υπέρ. Μπορούμε μαζί τις τρεις πρώτες τροπολογίες. Ωραία. Ποιοι είναι υπέρ τις πρώτες 2 και 3. Κατά. Αποχές εγκρίθηκαν. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 13-12. Τροπολογία 12 τώρα. Και 13 μαζί. Ωραία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Κατά τμήματα τώρα ψηφοφορία στη 14. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Α, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίθηκε. 16, 9 και καμία αποχή. Στη συνέχεια 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα, Επιτροπή Λίμπε. Λίμπε 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο τροποποιημένο. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας τη 22 υπέρ, ένας κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια. Και συνεχίζουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι στη Γραμματεία για τη βοήθειά της, γιατί πραγματικά έχουμε πολλά να ψηφίσουμε και είχαν πολλά να προετοιμάσουν. So, now Λοιπόν, τώρα. Ερχόμαστε στην απαλλαγή των οργανισμών. Και ξεκινάμε Έχουμε την έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018. Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος. Η συγητή είναι ο κύριο Τσαρνέσκι. Θέλετε μήπως το λόγο κύριε Τσαρνέσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω το προσωπικό και όλους όσοι βοήθησαν. Πολύ καλή δουλειά και να σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, τροπολογία αριθμό 1. Α, μία, ε, η πρώτη και η δεύτερη μαζί. Τροπολογίες 1 και 2. Και 3, αν θέλετε, ναι. Ωραία. 1, 2 και 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. 4 υπέρ. Τροπολογία 4, ναι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6, υπέρ, Πανέβασε εκτός μικροφώνου. 6 και 7 μαζί. Γίνεται. Όχι. Ωραία. Τροπολογία Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Καταπίπτει. Και η 9 καταπίπτει. Φτάνουμε στη 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω θα ελέγξουμε όμως. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα ναι, ψηφίσατε όλοι. Ωραία, πέρασε τις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 12 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 13. 13, 14 και 15 μαζί γίνεται. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18, 19 και 20 μαζί. Γίνεται. Όχι. Ωραία. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Θα δούμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε.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 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρεις τροπολογίες Λάρα Βόλτερς μαζί, συμφωνείτε. Υπέρ παρακαλώ και των τριών, κατά, αποχές εγκρίνονται. 34 καταπίπτει, 35 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να έλεξουμε. Ωραία. Αν θέλετε να επαληθεύσουμε, ευχαρίστως. 37, παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρασε. 18-4. 38 καταπίπτει. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Υπέρ τη 41. 41 με 44 υπέρ. 41 με 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Καταπίπτει 43. 45 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία. Αριθμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για να δούμε 49, 50 και 51 μαζί, ναι. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 52, 53 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 54 και 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 και 59 μαζί υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίνονται 58 και 59. Η 60 καταπίπτει. Η 61 επίσης. 62 τώρα. Και 63 μαζί. Υπέρ. 62 και 63. Κατά. Αποχές. Έγκρινονται. Η 64 καταπίπτει. 65 και 66 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 67 καταπίπτει. 68 και 69 μαζί τώρα. Ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 70 και 71 τώρα. Μέχρι την 74? Όχι. 70 και 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Να ελέγξουμε. Ε, εντάξει, βεβαίως. Ελέγχουμε. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Μαρία πάλι έχασες νομίζω. 16-7-1. Σαστέρ. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια περνάμε στις τροπολογίες της ΕΜΠΛ. ΕΜΠΛ 10 Έμπλ 11. Μια στιγμή, μια στιγμή. 10 και 11 καταρχήν. Υπέρ. Υπέρ 10 και 11 της Apple. Κατά. Εγκρίθηκαν. 12 και 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Και τώρα τις Λίμπε. Η 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεπώς, ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας, 21 ψηφί υπέρ, 3 κατά και καμία αποχή. Και περνάμε τώρα στις επιμέρους οργανισμούς με τρεις εισηγητές, Τζανέτσκι, Μπρουζίνσκι και Λιγκούλκο από το ECR. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα για το 1 Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, λέει πρόεδρο. Λοιπόν, η υπηρεσία για τη για τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, ε, τροπολογία 1 που είναι ίδια με την τροπολογία 2, για την απαλλαγή, χορήγηση απαλλαγή δηλαδή, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση για την απαλλαγή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 19, 3, καμία αποχή. Πολύ ωραία. Και τώρα πάμε απευθείας στην τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά να το ελέγξουμε παρακαλώ πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 14-2 8, συγγνώμη. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Όχι καταπίπτει. 9 καταπίπτει. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο επί του συνόλου όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 20 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή και πάμε τώρα στο Μπέρεκ ε, που είναι το γραφείο για το όργανο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για κοινωνικέ επικοινωνίε Μπέρεκ, υπέρ για το 1 και το 2, κατά Αποχέ εγκρίνεται. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η απόφαση. Τώρα επιβεβαιώνουμε την απόφαση τη απαλλαγή. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Είκοσι 3 και καμία αποχή. Και τώρα έχουμε την τροπολογία 4 υπέρ. Α, όχι. Τροπολογία 4, ναι, υπέρ. Κατά. Αποχή, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 καταπίπτει 10 10 και 6 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 Καταπίπτει 13. 14 και 15 από κοινού όχι. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κα... έχουμε κάποια ιδιαίτερη φιλία και συμμαχία κατά αποχή εγκρίνεται. Λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία τώρα επί του συνόλου του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ 3, 3 κατά καμία αποχή και τώρα περνάμε στο μεταφραστικό κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία 1 και 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα νομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλλον όχι ακόμα. να ψηφίσουν και οι τελευταίοι παρακαλώ. Κάποιος λείπει ακόμα. Μάλιστα, πέρας ψηφοφορίας, 20 υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές. Και τώρα περνάμε... Α, 0 αποχές, συγγνώμη, δεν υπάρχουν αποχές. Και τώρα τροπολογία 4 και 5 από κοινού, αν δεν έχετε αντίρρηση, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 και 7 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 και 10 9, 10 και 11 και 12 και 13 9, 10, 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μαρία εδώ έχουμε ιδιαίτερη φιλία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα πάμε στην κουλτ 327 υπέρ κατά 3 έως 7 μάλλον, εγκρίνονται. Και τώρα ε, ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου, άρχεται ψηφοφορία. «23 υπέρ, καμία ψηφοκατά και τώρα πάμε στην απαλλαγή για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τροπολογία 1 και 2, υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 υπέρ. Τροπολογία 4 και 5 από κοινού, αν δεν έχετε αντίρρηση, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα 6 και 7 6 μάλλον καλύτερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μαρία είσαι μόνη λυπάμαι Είσαι το άτυχο κορίτσι σήμερα. 9. Εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία δεν φαίνεται να υπάρχει αντίρρηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 13 υπέρ, 7 κατά, 3 αποχές. 10 και 11 από κοινού υπέρ. Όχι, όχι, δεν συμφωνείτε. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά θα δούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 7 υπέρ, 9 κατά, 7 αποχές. Ενδιαφέρον. 12 υπέρ, κατά. Πάλι θα πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά να δούμε. Πέρας ψηφοφορίας. 13 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται. 13 και 14 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 15 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται Άρχεται ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Ναι, 13 υπέρ, 9 κατά, έχετε δίκιο. 16 και 17, όχι 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 18, διότι 17 καταπίπτει. 18 ε, και 19, όχι, 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη φιλία που γεννιέται. Να δούμε την, από 3 έως 5 ή από 3 έως 12 της ΕΝΠΟΛ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία επί του κειμένου όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία. Όλα υπερψηφίστηκαν τη Επιτροπή Απασχόληση. Λοιπόν, πέρα τη ψηφοφορία, 19 υπέρ, 3, 3 κατά, καμία αποχή. Και τώρα σε πολ. Τροπολογία 1, 2 και 3. Υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνονται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απαλλαγή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 21 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Και τώρα έχουμε την τροπολογία, τροπολογίες 6 και 7. Υπέρ, υπέρ τις 6 και τις 7, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα 8 και 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 10 υπέρ, κατά αποχές να το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία για τη 10 πέρας ψηφοφορίας 11 υπέρ εγκρίνεται 8 κατά 4 αποχές 11 εδώ έχουμε προφορική τροπολογία έχει κανείς αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν επί της 11 υπέρ κατά αποχές ενδιαφέρον. Θα πρέπει και αυτό να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας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 από κοινού. Ναι, εντάξει, ναι, 20-21, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε τώρα. Έχουμε μερικώς καλύψει την παράγραφο 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μόνο Είχαμε χωρομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Είκοσι υπέρ, τρεις κατά, καμία αποχή. Είσαστε σκληροί και, και εξαιρετικά πειθαρχημένοι. Συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα στην ΕΑΣΑ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, παράγραφος 1, τροπολογία 1 και 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ονομαστική ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής υπέρ μάλλον άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 20 υπέρ 2 κατά μία αποχή τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 και 7 6 και 7 από κοινού ωραία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 και 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 10 και 11. 10 και 11. Υπέρ. Όχι, μόνο τη 10. 10, 10. Υπέρ της 10. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε Μαρία δυστυχώς. 11. Υπέρ. Και 12 μαζί. Όχι. 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λοιπόν τραν 3 έως 9 τροπολογίες τραν 3 έως 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και τώρα να δούμε την 10 την 11 την 13 όχι τη 14 10 έως 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 14 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω να το επαληθεύσουμε βεβαίως πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 11-11 Δεν το περίμενα. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα επί του κειμένου στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε άρχιτη ψηφοφορία. Είκοσι υπέρ, δύο κατά, μία αποχή και τώρα πάμε στην ΕΑΣΟ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τροπολογίες 1, 2 και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση απαλλαγής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας 19 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Και πάμε στις τροπολογίες. Τροπολογία 7 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 και 9 καταπίπτουν και η 10 11 ποιος είναι υπέρ κατά θα πρέπει να το δούμε αυτό τώρα να το επαληθεύσουμε την ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας 10 υπέρ 13 κατά απορρίπτεται χωρίς αποχές 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15, 12 και 15 καταπίπτουν, μάλλον 14 καταπίπτουν, συγγνώμη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 και 17 καταπίπτουν 18 υπέρ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 23 23 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 κατά πίπτη 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 καταπίπτει 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 καταπίπτει, 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 πίπτη. 37 κατά πίπτη. 38 υπέρ. 3, κατά αποχές εγκρίνεται. 39 κατά πίπτη. 40 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 41 κατά καταπίπτει 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά α... αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 κατά πίπτη 49 και 50 από κοινού την έχετε αντίρρηση 49 πρώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Και τώρα περνάμε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 1, 2, 3. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα που επιβεβαιώνει την απόφαση απαλλαγής. άχρη ψηφοφορία. Λείπουν δύο. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 4 κατά και τώρα 5. Λάρα Βόλτερς, ε, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι να το ελέγξουμε να το ελέγξουμε ήταν λίγο αυτό 8 λοιπόν τροπολογία 8 Ωραία, πέρας ψηφοφορίας. 13 υπέρ, 7 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι έγκρινεται 10 υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται 12 καταπίπτη ή 11 καταπίπτη 13 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική α ποιος είναι υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 23 υπέρ κατά να το ελέγξουμε. Close the vote. 13 plus 10 minus no abstentions. Then 20... Εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην έκον αυτό ήθελα να πω 2-2-7 ή μάλλον 2-2-9 2 μέχρι συγγνώμη μέχρι 9 2 μέχρι 9 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται μετά έχουμε 12, 13, 16, 17 Εφικτό, ναι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της όπως τροποποιήθηκε άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 20 εναντί 3 και 0 αποχές. Πάμε στην ECDC, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. <laughs> Θέλει κανείς να πάει προς νερού του. Ναι. Θα το συζητήσουμε πρώτα, λέει. Very shortly come back, Thomas. Να έρθετε, Τόμας, πολύ γρήγορα. But... Maria, we need, they need a short break. It's really tough, but we are on our way. Yeah, it's fine. So Θα ήθελα να παρακαλέσω τα μέλη να επιστρέψουν. we are welcoming you. Λοιπόν, επιστρέψτε. Yes. Okay. ECDC. ECDC. Πάμε. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρ κατά αποχές εγκρινώνται ε, ονομαστική ψηφοφορία για την επικύρωση της απόφασης απαλλαγής. Ψηφίζουμε ακόμα ηλεκτρονικά. Πόσα μέλη έχουν μείνει εδώ. Νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε. 18 περμία μία κατά καμία αποχή. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αεγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται NV να ψηφίσουμε αν μπλοκ όλες τις MV ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματο στο σύνολό τη και άρχεται η ψηφοφορία ωραία πέρας ψηφοφορίας 20 υπέρ, μία κατά, καμία αποχή. Πάμε ΕΚΑ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, τροπολογίες 1 και 2. Ποιος είναι υπέρ? ΕΚΑ. ΕΚΑ. Τροπολογίες 1 και 2 του κυρίου Σεντοφσκή και Πέτρη Σαβαρβάμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται ονομαστική ψηφοφορία για την κύρωση της απόφασης απαλλαγής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 υπέρ, 2 κατά, 0 αποχές. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε. Πρέπει να βάλουμε μια κρυφή κάμερα. Ε. Υπέρ. Απέρα, συγγνώμη. 11. Υπέρ 10 κατά. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 και 9 μπορούμε ναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 κατά πεπτή 12 και 13 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 14 και 15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 εγκρίνονται. Οι 20 και 21 είναι ταυτόσιμες. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβη να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Unblock, ναι, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται όλες ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο, για το, πρώτο ψηφίσματος στο σύνολό τη. άρχεται η ψηφοφορία πέρας 19-2-2 0 2 κατά 0 αποχές Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τροπολογίες 1 και 2 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία για την κύρωση της απόφασης απαλλαγής. Άρχεται η ψηφοφορία. Εξακολουθεί να τρέχει η ψηφοφορία πέρας. 19 προς 2 και 0 αποχές. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να πάρουμε τις 6 και 7. 6 μόνο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 καταπίπτει 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11, 12 και 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται οι 11, 12 και 13, 14 και 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 16 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. έναρξη ψηφοφορίας λήξη 10 υπέρ 9 κατά 3 αποχές 17 υπέρ κατά η ίδια πλειοψηφία να ελέγξουμε ελέγχουμε λοιπόν την 17 Καλή προσπάθεια. Τώρα απορρίπτεται, Τόμας. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται, Μαρία. ένβι Να ψηφίσουμε unblock. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19-3 με αποχές. Η FCA, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλίας. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία που κυρώνει την απόφαση απαλλαγή υπέρ. Αν έρχεται ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας. 19, 3, 0 αποχές. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται 6 και 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 8 και 9. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα έχουμε την ΠΕΣ ε, μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί α, τις 7, 8, 9, 10, 11 και 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολο όπως τροποποιήθηκε άρχεται ψηφοφορία πέρας όχι Λείπουν δύο. Τζόζεφ. Πέρας. 19 υπέρ 3 κατά. Μηδέν αποχές. Εύσα, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία για την κύρωση της απόφασης απαλλαγής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 υπέρ, 3 κατά, 0 αποχές. Τροπολογίες 4 και 5. Και 6 μαζί. Όχι, 4 και 5. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνονται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές κάποιοι δεν, έβαλα, δεν ψήφισαν άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά Ο Τζόσεφ ε, δεν ψήφισε και πάλι είστε το θύμα μας σήμερα. 15-4-3. 7 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά δεν είμαι βέβαιη. Πέρας. εγκρίθηκαν 12 προς 9 θα ήταν λάθος 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ 9 και 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 11 καταπίπτει 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ 13 υπέρ Κατά. Να ελέγξουμε. Ένας λείπει. Ωραία. 13 υπέρ, 6 κατά εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί Renew είναι κατά. Να ξαναελέγξουμε την 14. Πέρας. 12 υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται 16 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 15 πίπτη. 17 υπέρ κατά να ελέγξουμε διότι οι πράσινοι προσπαθούν να βρουν ε, πόζα να πάρουν για φωτογραφία 17 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 18 ποιος είναι υπέρ Κατά. Να ελέγξουμε. Αλλά νομίζω ότι εγκρίνεται. 19. Ποιος δεν ψήφισε. Ωραία. Εγκρίνεται. 11 υπέρ 10 κατά. Εγκρίνεται. 19 κατά καταπίπτει. 20. Ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε όλες τις έμβοι μαζί ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό τη. Όπω τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 έναντι 3 0. Συνεχίζουμε τώρα και πηγαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ποιοι είναι υπέρ των τροπολογιών 1 και 2. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για να επιβεβαιώσουμε την απόφαση από αλλαγή. Ψηφίζουμε. «18 υπέρ, 4 κατά και καμία αποχή». Τροπολογία αριθμός 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 και 8 μαζί. Υπέρ τη 7 μόνο. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, Α, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίφθηκε 10-12. Τροπολογία 10. Εδώ έχουμε προφορική τροποποίηση. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροποποίηση. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε τότε με την προφορική τροποποίηση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Σηκώνετε τα χέρια παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται γιατί οι πράσινοι απέχουν. 11 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 καταπίπτει. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογίες γυναικών, της Επιτροπής Γυναικών. Παράγραφος 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Παράγραφος 2 της Επιτροπής Γυναικών. Δώδεκα επτά. Τώρα για οι υπόλοιπε των γυναικών, υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα του συνόλου του κειμένου τροποποιημένου. Μπορείτε να ψηφίσετε. 18 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Και συνεχίζουμε με την ΑΙΟΠΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Τροπολογίες 1 και 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα που επιβεβαιώνει την απόφαση για την απαλλαγή. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 17 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Τροπολογία αριθμός 3. Υπέρ. <clears throat> κατά. Απορρίφθηκε. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 και 7 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 8 και 9. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνονται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, έχουμε τις τροπολογίες της Οικονομικής Επιτροπής. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Ωραία, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα επί του τροποποιημένου κειμένου. Ψηφίστε παρακαλώ. Δεκαεννέα υπέρ, δύο κατά και μία αποχή. Και ερχόμαστε τώρα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Τροπολογίες 1 και 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκαν. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα που βεβαιώνει την απόφαση απαλλαγής. Μπορείτε να ψηφίσετε. «19 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή». Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνατε. 5 και 6, 5 μόνο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 και 8. Μαζί γίνεται, ωραία. 7 και 8 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 9 και 10. 9 και 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 και 13 <clears throat> υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 14 και 15, 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα στο τροποποιημένο κείμενο μπορείτε να ψηφίσετε. 19 υπέρ, 3 κατά. Έμα τώρα. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για την επιβεβαίωση της απόφασης απαλλαγής. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ποιος το ψήφισε, Τζόσεφ, εσύ πάλι. Είμαστε όλοι υπέρ, ναι. Καταλαβαίνω. 18 υπέρ, 3 κατά. Καμία αποχή. Τροπολογία 4 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6. Να ελέγξουμε. Ναι, βεβαίω. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. 7-7-6 είναι το αποτέλεσμα. Το λήξαμε. 7-7, άρα απορρίπτεται. 6 τώρα, τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 και 8, όχι, 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ, 8 και 9 Ωραία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 10 καταπίπτει. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13, 14, 13 και 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 16 τώρα. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 17 και 18 μαζί και τη 19 μαζί όχι 17-18 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 και 20, όχι, 20 μόνο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 και 25. 24 μόνο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί όλες τις τροπολογίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Όλες τις έμβε μαζί λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και τώρα το σύνολο του κειμένου τροποποιημένο. Ψηφίστε παρακαλώ με ονομαστική ψηφοφορία. 20 υπέρ, 3 κατά. Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Τροπολογίες 1, 2 και 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία και επιβεβαίωση της απόφασης απαλλαγής. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 ε, υπέρ, 2 κατά. Καμία αποχή. Τροπολογία τώρα αριθμός 6. 7 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 και 10 μαζί υπέρ κατά Α, μόνο την 9 θέλετε. Ωραία, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 και 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 15 και 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 17, 18 και 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 20 και 21, 20 μόνο. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα τροπολογίες της ΛΥΜΠΕ, τις δύο που έχουμε μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του τροποποιημένου κειμένου. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 2 κατά. Καθόλου αποχές. Και περνάμε τώρα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Τροπολογίες 1 και 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για την επιβεβαίωση της απόφασης απαλλαγής. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. 20 υπέρ, 2 κατά, ε, καμία αποχή. Τροπολογία αριθμός 4 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 6 και 7 και 8 6-7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 και 10 όχι 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 πίπτη, 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, έχουμε μεταφορές. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί όλες τις τροπολογικές επιτροπές μεταφορών. Καλώς. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. 20 υπέρ, 3 κατά. Καμία αποχή. Συνεχίζουμε την ενίζα. Οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, τροπολογίε 1 και 2 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία για την επιβεβαίωση της απόφασης απαλλαγής. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. 20 υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Τροπολογία αριθμός 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τέλος της ψηφοφορίας. 12 υπέρ, 8 κατά και 3 αποχές. Τροπολογία αριθμός 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπάρχει προφορική τροποποίηση εδώ. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική. Όχι. Συνεπώς, τότε ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ναι, ναι. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά... 13 υπέρ, 7 κατά. Δίκιο είχατε. 7 και 8 τώρα. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται. Να ήταν οι 7 και 9. Ε, οι 8 καταπίπτει, 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα με ονομαστική ψηφοφορία το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε. Τέλος. 21 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Και συνεχίζουμε και περνάμε τώρα στον Οργανισμό Σιδηροδρόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρ, κατά. Εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για την επιβεβαίωση της απόφασης. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. 19 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Τροπολογία αριθμός 6 τώρα. Α, και η 6 έχει αποσυρθεί, οπότε 7, 8 και 9 μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνονται, αλλά θα δούμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 13 ψήφοι υπέρ, 9 κατά και μία αποχή. Τροπολογία αριθμός 10 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Να ελέγξουμε τη 10. Κύριε Κούς, ψηφίσατε. Ωραία. 12 υπέρ, 8 κατά και 3 αποχές. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 και 16 υπέρ 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε η ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. 10 υπέρ, 12 κατά και μία αποχή. Απορρίφθηκε. 18 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί το όλες τις τροπολογίες της Επιτροπής Μεταφορών. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Και εγκρίθηκαν. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε στο σύνολό του. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. 20 υπέρ, 3 κατά. ΕΣΜΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, τροπολογίες 1 και 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία για την επιβεβαίωση της απόφασης απαλλαγής. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. 18 υπέρ, 2 κατά, 1 αποχή. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, Εγκρίνατε νομίζω, αλλά θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος. 11 υπέρ, 9 κατά μία αποχή. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται νομίζω. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται νομίζω. 11 και 12 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 13 και 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 15 καταπίπτει. 16 και 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 18 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέλος, απορρίφθηκε. 19 λοιπόν τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20, υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά παληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. εγκρίθηκε. 11-10. Τώρα, έχουμε όλες τις τροπολογίες της Οικονομικής Επιτροπής. Γίνεται. Ωραία. Υπέρ, παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορία 20 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή. Και τώρα ETF, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ονομαστική ψηφοφορία πρώτα, άρχιτη ψηφοφορία, Πέρας ψηφοφορίας 20 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Τροπολογία 1 και 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι δεν εγκρίνεται απορρίπτεται εννοώ απορρίπτεται εννοώ να το ελέγξουμε πάντως απορρίπτεται νομίζω Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα όλες τις τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και τώρα η ονομαστική ψηφοφορία ε, επί του συνόλου το κείμενο που τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, 20 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή και τώρα η EU-LISA. Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής Μεγάλης Κλίμακας στο χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Τροπολογίες 1, 2, 3 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τώρα επί της επιβεβαίωσης της απόφασης απαλλαγής υπέρ, ή μάλλον άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, 20 υπέρ, 3 κατά, μία, καμία αποχή, 4 και 5 καταπίπτουν, τροπολογία 6, 7, 8, 9 από κοινού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται να ψηφίσουμε από κοινού 10 και 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 12 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 13 κατά πίπτη 14 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 καταπίπτει, 17 καταπίπτει, 18 και 19 από κοινού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 και 21 καταπίπτουν, 22, 23 και 24 από κοινού. Όχι, 22, 23 και 24, ναι. Όχι, όχι, 22, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 και 24 τώρα από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε επί της 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα 26 κατά πίπτη, Ναι, το 20 δεν εγκρίθηκε όμως, οπότε πρέπει να ψηφίσουμε επί της 26. Υπέρ της 26, κατά αποχές εγκρίνεται. 27-28 από κοινού, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ε, τις τροπολογίες της ΛΥΜΠΕ όλες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και ψηφίζουμε τώρα επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε άχετε ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ 3 κατά 0 αποχές και τώρα EU OSA, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Τροπολογίες 1, 2, 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση απαλλαγής. Άρχεται η ψηφοφορία. Να περιμένουμε και την Καταλίνα. Μικρή αλλαγή. Σας περιμένουμε, μην ανησυχείτε. Πέρας ψηφοφορίας, 22 υπέρ, 3 κατά. Χαιρετούμε τον Ολιβιέ. Πολύ πειθαρχημένο σήμερα, ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στην τροπολογίε στις τροπολογίες 6 και 7. Ψηφίζουμε για την 6, 7 και την 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 και 12. Μόνο 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες της ΕΜΠΛ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και τώρα ψηφίζουμε ονομαστικά επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκα η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 20 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή και τώρα πάμε στην ESA, ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ, τροπολογίες 1 και 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση απαλλαγή υπέρ ή μάλλον όχι. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 19 υπέρ 3 κατά καμία αποχή τροπολογίες 4, 5 και 6 4 και 5 4 και 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ 6 και 7 από κοινού ωραία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία ε, επί του κειμένου όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Eurofund, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνδικών Διαβίωσης και Εργασίας. Τροπολογία 1 και 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση απαλλαγής. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας 20 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 4 και 5. Όχι, 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας 11 υπέρ 6 κατά 5 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 6 και 7. Όχι, όχι. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 και 8 αν θέλετε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα όλες τις τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ 3 κατά Eurojust τώρα Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας τροπολογίες 1, 2 και 3 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ονομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση απαλλαγή. άρχεται ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας 20 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή και τώρα πάμε στην τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 και 8, όχι. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα οι τροπολογίες της ε, ΛΥΜΠΕ 3, 6 και 4, 6 και 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τραποποιήθηκε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 2 κατά. Και τώρα περνάμε στην Ευρωπόλ, Οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συνεργασία στον τομέα τη επιβολή του νόμου. Τροπολογίε 1, 2 και 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση απαλλαγή. Υπέρ. Ή μάλλον άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. ψηφοφορια δίκιο. Είμαστε κοντά στο τέλος. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί πάντως από την πειθαρχία όλων εδώ. Πάμε... Ε, ναι, 21 υπέρ ψήφι. 2 κατά καμία αποχή, τροπολογία 4 και 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 6, τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 7 και 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Εντάξει, νομίζω πάντως ότι απορρίπτεται. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 11 υπέρ 12 κατά. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα την τροπολογία 11. Εδώ έχουμε προφορική τροπολογία. Έχει κανείς αντίρρηση? Όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπορούμε είναι καταπίπτει. η Επόμενη 14 και 15 από κοινού, όχι. 14 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 12 υπέρ, 7 κατά 4 αποχές, εγκρίνεται 15 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 και 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 καταπίπτει. Και τώρα 19 και 20. Όχι. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συνεχίζεται αυτή η συμμαχία η ειδική δεκαετία υπέρ κατά αποχές Άμυρη Μαρία εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, ψηφίζουμε και τις δύο τροπολογίες της ΛΥΜΠΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ψηφίζουμε επί του του κειμένου όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας, 21 ψήφι υπέρ, 1 κατά, 1 αποχή. Και τώρα πάμε στην FRA, ο Οργανισμός Θεμελιδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αντίστροφη μέτρηση, 1, 2, 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται ονομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση απαλλαγή, άρχεται ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, 18 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή και τώρα πάμε στην τροπολογία 6 και 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται και οι δύο. 8 και 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εδώ θα πρέπει να το ελέγξουμε μάλλον τροπολογία 12 άρχεται ψηφοφορία αυτή τη φορά Γιώζεφ πρέπει να, να υπερψηφίσεις. Απορρίπτεται. 10 υπέρ 11 κατά 2 αποχές. Τροπολογία 13. Προφορική τροπολογία. Αν δεν έχει κανείς αντίρρηση, ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 και 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 κατά πίπτη, 18 και 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα όλες τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ από κοινού παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 8 ψήφι. υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Frontex, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Νοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. 1, 2, 3. Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ομαστική ψηφοφορία που επιβεβαιώνει την απόφαση απαλλαγή. Άρχεται η ψηφοφορία. Close. Πέρας. 19, 3 και μία αποχή. Έχουμε την τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 9, 10, 11 όλες καταπίπτουν 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γλωσσικές τροπολογίες 6 και 17 16 η ειδική φιλία πρέπει να συνεχίσει υπέρ κατά εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές φτωχή Μαρία Άμερ Μαρία ε, εγκρίθηκε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε αλλά νομίζω ότι να ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρασε 11, 9, 3, εγκρίνεται. Τέλεια Μαρία, όλα άψογα. 21 και 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται και τα δύο. με δεν αλλάζει η πλειοψηφία. Αν δεν έχετε αντίρρηση, αφού δεν αλλάζει. 23. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Εγκρίνεται νομίζω. Αλλά να ελέγξουμε. Να ελέγχουμε την 23 πέρας ψηφοφορίας 12-10 εγκρίνεται και μία αποχή 24-25 24 και 25 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 και 27 υπέρ κατά αποχές εγκρινώνται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ 35 υπέρ κατά αποχές και οι δύο εγκρινώνται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 καταπίπτει 34 υπέρ κατά αποχές γκρινέται, η φιλία συνεχίζεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές η Μαρία απορριφθήκε τώρα αλλά η Εγκρίθηκε η τροπολογία λίμπε. Νομίζω ότι ψηφίσαμε όλες ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τώρα έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Πέρας 19-2-1 τελευταίος οργανισμός. Κοινέ επιχειρήσει, αλλά δεν τόσε τόσο πολλέ. Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS ένα και δύο. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την κύρωση της απόφασης απαλλαγής. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε. Ψηφίστε ακόμα. Πέρας. 21, 1 και 0. Τροπολογίες 4 και 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρινώνται 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 7 και 8. 7 και 9 λέγεται στην αίθουσα. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 και 8. Όχι. Η 8 καταπίπτει. 9 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. 8 καταπίπτει. 10. 11 υπέρ κατά αποχές 10 και 11 εγκρίνονται 12 υπέρ κατά αποχές Άμυρη Μαρία εγκρίνεται ονομαστική ψηφοφορία για το πρόταση ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε 21-2 συγχαρητήρια στον κύριο Τζαρνέτσκι, στον κύριο Λεγκούτκο και Μπουτζίνσκι. Τώρα έχουμε τις κοινέ επιχειρήσεις. Οι τελευταίες οκτώ κοινέ επιχειρήσεις. Η συγγετής ε, είναι ο κύριος και Θέλετε το λόγο. Shortly, thank you much indeed. Εν συντομία σας ευχαριστώ όλους. So, we thank Όχι, εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν τόσο εξαίρετος συγγετής. Ευχαριστούμε πολύ. Τροπολογία 1 για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση απόφασης απαλλαγής στο σύνολό της όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται ψηφοφορία, ψηφίστε, πέρας. Δεκαεννέα δύο μηδέν. Πάμε τώρα στις τροπολογίες. Δύο υπέρ κατά να ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Πέρας. Απορρίπτεται, σαφώς. Τροπολογία 3, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά Α, να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας 10, 9, 2. 7, 8. 7 και 8. 7 και 8. Θα ήταν υπερβολικά πολύ γκραπίνη και Ζεντόφσκι σε μία ψήφο απίστευτο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται χωρίς εποχές, ε, ονομαστική ψηφοφορία. Για το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρας. 20 εναντί μίας. Ε, clean Sky, αεροναυτική και περιβάλλον. Μ' αρέσει αυτή την επιχείρηση. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση απαλλαγής πέρας 22 και έχουμε τώρα μια ψηφοφορία για την τροπολογία 2 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές, σας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Το ελέγχουμε. 4. Υπέρ. 4 και 5. Ωραία, περ, κατά αποχές εγκρίνεται 6 και 7 6 και 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 και 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται να τις ψηφίσουμε όλες μαζί, τις τροπολογίες Τραν. Ωραία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Πάμε τώρα στην ονομαστική ψηφοφορία για το νέο ψήφισμα αυτό που τροποποιήθηκε. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 εναντί 2 και 0. Συνεχίζουμε με το Excel, την κοινή επιχείρηση, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Τροπολογία αριθμός 2 και 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 5 και 4 υπέρ, κα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 και 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 και 9 υπέρ κατά 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε. 19-2. Συνεχίζουμε. Κυψέλη καυσίμου και υδρογόνο 2. Τροπολογία αριθμό 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή. Τέλος της ψηφοφορίας. 19-2. Παράγραφος 11, τροπολογίες 2 και 3. Γίνεται μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 4 και 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 6 και 7. 6 μόνο. Υπέρ, κατά, αποχές, θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίφθηκε σαφώς 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα ε, για το σύνολο. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 19 υπέρ 2 κατά καμία αποχή. Και ερχόμαστε στο IMA που είναι πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα. Τροπολίγα αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, Ονομαστική, Ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Ξέρω ότι είναι αργά και είναι δύσκολο για όλους. Ωραία, τέλος. 19 υπέρ. Καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Τροπολογίες 3 και 4. Μαρία και Τόμας μαζί σε μία ψηφοφορία. Δεν γίνεται. Ωραία. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 και 5 μαζί. Όχι. 4 μόνο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γκρίθηκα ο με τη βοήθεια της Μαρία. Ωραία, 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 και 7 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 8 και 9 υπέρ, κατά άποχες εγκρίνονται. 10 και 11, όχι, μόνο 10 υπέρ, κατά άποχες απορρίπτεται. 11 και 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 13 και 14 υπέρ των 13 και 14 κατά αποχές εγκρίνονται 15 και 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 17 και 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Αποτέλεσμα 20 υπέρ, ε, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Σύνδειξη. Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύνδειξης. Ήτερ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Σαφές. Τώρα σηκώστε τα χέρια. Αποχές. εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για την απαλλαγή. Ψηφίστε παρακαλώ. «15 υπέρ, 6 κατά και μία αποχή». Τώρα, ψηφίζουμε. Παράγραφος 5, τροπολογία αριθμός 2. 2 και 3 μαζί γίνεται. Ωραία. 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τέσσερα καταπίπτει. Πέντε, λοιπόν υπέρ. Μαρία, η τροπολογία σου καταπίπτει. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Καταπίπτης, είπε ο πρόεδρος. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μισελ 7 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Τώρα έχουμε την 8 σε δύο τμήματα Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα υπέρ έχει αποσυρθεί το δεύτερο τμήμα, ναι. Σωστά, 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 καταπίπτει. 11 και 12 υπέρ 11 και 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 και 14 όχι, 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, Όλα είναι εντάξει στο τέλος. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18-19. 18 και 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 καταπίπτει. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για το σύνολο του κειμένου που τροποποιήθηκε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Σέζαρ τώρα, κοινή επιχείρηση. Τροπολογία 1, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή υπέρ λέει η πρόεδρος. Ανοίγει, αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 19 υπέρ 3 κατά καμία αποχή. Τροπολογίες τώρα. Μπορούμε 2 και 3 μαζί. Ωραία, υπέρ 2 και 3. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 4 και 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 6 και 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 8 και 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 10 και 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται Απορρίπτεται. 13 και 14. Μαζί. Όχι, 13 μόνο. Υπέρ. Κατά. Τι θέλετε να λέξουμε. Την 12. Ωραία. Ελέγχουμε. Παληθεύουμε ηλεκτρονικά. Την 12. Ο Τόμας δεν πιστεύει ότι έχασε. Γι' αυτό. 11-11. Έχει δίκιο. Rejected. Απορρίπτεται. 13. Και 14. Όχι, ωραία. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες τραν, όλες μαζί. Ωραία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Τέλος της ψηφοφορίας. 19 υπέρ 3 κατά καμία εποχή. Shift to Rail, κοινή επιχείρηση. Είναι η τελευταία μας ψηφοφορία αυτή. Ωραία. Συνεπώς, τροπολογία αριθμός 1, υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή τώρα, υπέρ. Ψηφίζουμε βέβαια ηλεκτρονικά. Εντάξει, ψηφίσατε όλοι πέρας. 19 υπέρ, 2 κατά. Καμία αποχή. Τροπολογία αριθμό 2 και 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 4 και 5, όχι. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 και 8 και ναι, όχι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Όλες οι τροπολογίες τραν τώρα μαζί. Μαζί. να ξαναψηφίσουμε, αλλά ψηφίσαμε και τις τρεις. Τροπολογία 9. Ξαναψηφίζουμε, αν και την ψηφίσαμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και πάλι. Τραν τώρα. Οι τροπολογίες τραν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Και τώρα η τελευταία ονομαστική ψηφοφορία, η τελευταία μας απαλλαγή για το 18, μπορείτε να ψηφίσετε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια σε όλους. Τα καταφέραμε. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την πειθαρχία. Sorry, sorry, just. Tomorrow continue, we continue at 9 for the coordinated... Tomorrow we continue at 9 at... Αύριο στις 9 με τους συντονιστές και ανοιχτή η συνεδρίαση από τις 10.30. Ευχαριστώ πολύ. 9 the coordinators. At... Στις 9 οι συντονιστές. 10.30 η κανονική συνεδρίαση. Ευχαριστώ για την πειθαρχία που επιδείξατε. Είσαστε μια καταπληκτική επιτροπή.